και να αναπτυχθεί ως ένα σώμα υπέρ της ειρήνης και της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό όσον αφορά τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ. Έχω να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Από τους εισελιστές μου ζητήθηκε ορισμός σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Ο κατάλογος θα είναι στα πρακτικά τη συνεδρίαση αυτή Εφόσον δεν έχει υπάρξει καμία παρατήρηση μέχρι να εγκριθούν τα πρακτικά, οι ορισμοί αυτοί θεωρούνται εγκεκριμένοι. Και περνάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Είναι ο κοινωνικό πυλώνα τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Πρόκειται για δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώ, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον πρόεδρο Μπαρόζο συλλογικά εργάζεται για την προετοιμασία μίας πρότασης που θα ενδυναμώσει τον κοινωνικό πυλώνα της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Πρόκειται για μέτρα που αρμόζουν για την καλύτερη λειτουργία της ε, ζώνης ευρώ αλλά και για την προετοιμασία της κοινωνικής ατζέντα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Εν ώψη της υψηλής ανεργίας και της ύφεση σε πολλά τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στα πλαίσια της εντολής τους να εργαστούν. Το κάθε κρατός μέλος μεμονωμένα αλλά και από κοινού για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Στοχεύουμε την επαναφορά της ανάπτυξης, την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όλες οι πολιτικές μας έχουν αυτόν τον σκοπό. Η δημοσιονομική πολιτική για την δημοσιονομική εξυγένση των ε, δημόσιων οικονομικών κάτι που έχει ξεκινήσει και φυσικά θα πρέπει να συνεχιστεί με αυξημένους ρυθμούς. Θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν οι προσπάθειες έτσι ώστε με έντονο τρόπο να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα ή να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές οι κοινωνικές αυτές πολιτικές με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Να δοθούν εγγυήσει. Γι' αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, θα πρέπει να βρούμε τρόπους για καλύτερη ολοκλήρωση αυτής της κοινωνικής πτυχής στην παρούσα οικονομική διακυβέρνηση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει καλύτερη επαγρύπνηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όλων των πρωτοβουλειών που έχουν σαν σκοπό κοινωνικά μέτρα και βεβαίως χρειάζεται εις βάθος μεταρρύθμιση, ανάλυση των κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας με σκοπό να βρούμε τις αρνητικές επιπτώσεις και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται συντονισμένες πολιτικές έτσι ώστε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι πολιτικές αυτές που θα μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα όσον αφορά τα εργαλεία και τα μέσα που διαθέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ελαφρύνουμε τα κοινωνικά προβλήματα και τις δυσκολίες σε κάποιες χώρες πιο συγκεκριμένα. Η διασφάλιση της στήριξης μέσω των κοινωνικών ταμείων για μέτρα που θα καταπολεμήσουν την φτώχεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εδώ έχουμε επίσης και τα διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία θα πρέπει σαφώς να καταπολεμήσουν επίσης αυτά τα κοινωνικά προβλήματα. Η αξιολόγηση, ο αναπρογραμματισμός, η κατεύθυνση σε νέους τομείς κάποιας οικονομικής βοήθειας που προβλέπεται για άλλους τομείς είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Επίσης, η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης προϋποθέτει την ενσωμάτωση μιας πολιτικής που αφορά την αγορά εργασίας και αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την σωστή ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, της εσωτερικής αγοράς της Ευρώπης έτσι ώστε να φτάσουμε σε καλύτερα επίπεδα απασχολησιμότητας. Η κινητικότητα, η ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ευρώπης θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων, κάτι που πραγματικά μαστίζει συγκεκριμένα κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο θα πρέπει να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία μας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, χρειάζεται στενότερη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων σε αυτήν την πολιτική είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει, είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής και αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αξιοπιστία των πολιτικών μας και θα υπάρξει και καλύτερος πολιτικός συντονισμός. Είναι ζωτική σημασία λοιπόν να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Εξ ονόματος των ε, πολιτικών ομάδων του ΕΛΚ, ο κύριος Μάννα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε. Αναφερθήκατε πολύ σωστά στο γεγονός ότι η ύφεση θα πρέπει να μας οδηγήσει σε κοινέ λύσεις, κοινέ αντιμετωπίσεις και ότι δεν μπορεί τα κράτη-μέλη να ανακοινώνουν τα εθνικά τους μέτρα και την πολιτική τους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη ανάλυση των επιπτώσεων. Η κοινοτική λοιπόν συνεργασία θα πρέπει να ενδυματωθεί και θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές συζητήσεις πριν ανακοινωθούν εθνικά μέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επίσης πώς λειτουργεί η ενιαία αγορά, η εσωτερική αγορά. Και Σήμερα έχουμε δημιουργήσει βεβαίως τις προϋποθέσεις για ένα σταθερό ευρωπαϊκό νόμισμα. Πρέπει να, δημιουργηθούμε, να δημιουργηθούν συγγνώμη, προϋποθέσεις για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις. Η βιωσιμότητα της οικονομίας, η χρηματοδότηση υποδομών, αλλά και συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση εάν η οικονομική, νομισματική και κοινωνική πολιτική δεν στηρίζονται σε τρεις σταθερές βάσεις. Θα πρέπει στο μέλλον να ξεπεράσουμε την αντίφαση μεταξύ λιτότητας, εξοικονόμησης, περιορισμού των δαπανών και ανάπτυξης. Και αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε όλα τα κράτη-μέλη χρειάζεται η μείωση του δημόσιου ελλείμματος σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίως σήμερα είδαμε πολλοί επίπονα μέτρα να έχουν ληφθεί. Εξοικονομήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά που εξοικονομούνται για τομείς που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη, για επενδύσεις που στο μέλλον θα φέρουν θετικά αποτελέσματα. Οι πολίτες της Ευρώπης σήμερα βρίσκονται πολλές φορές σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση με μη μόνιμες θέσεις απασχόλησης και πολύ κοντά στο όριο της φτώχειας. Η ανεργία των νέων απαιτεί μία ορθή αντιμετώπιση και απάντηση από μέρους μας. Θα πρέπει να περιορίσουμε την ε, πολιτική μας από τις αρνητικές επιπτώσεις που δυστυχώς συνεχίζει να έχει. Έχουμε σήμερα διάφορες δυνατότητες αντιμετώπισης αυτών των οικονομικών φαινομένων όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα κοινωνικά ταμεία που πολλές φορές δεν χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται βιώσιμη αντιμετώπιση, προληπτική κοινωνική πολιτική σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει οι πολίτες της Ευρώπης να συμμετάσχουν με κατάρτιση, με εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Μάν. Η κυρία Μπέρες τώρα παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. 14 Μαρτίου μου αναλάβατε την επιστολή να ετοιμάσετε ένα χάρτη πορεία για την ολοκλήρωση τη ΟΝΕ από κοινού με τον πρόεδρο Φαν Ο χάρτη αυτό πορεία συμπεριλαμβάνει τέσσερι διαστάσει. Το Σώμα των Επιτρόπων κατέληξε σε δύο προτάσει υπό τη δικιά σα ευθύνη και αρνείται να μας δώσει το κείμενο το που εμείς περιμένουμε για τον κοινωνικό τομέα. Αλλά συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει. Είναι μια κατάσταση η οποία αποδεικνύει την αποτυχία της δικιάς σας πολιτική και η σιωπή του Σώματος των Επιτρόπων όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ είναι κάτι το οποίο δείχνει και την αποτυχία της Προεδρίας του κύριου Μπαρόσο. Δεν θα πετύχετε τίποτα. Δεν θα μπορέσετε να μας βγάλετε από την ανισορροπία που βρισκόμαστε, που δεν είναι μακροοικονομική. Δεν θα τα καταφέρετε αν δεν δείτε τι γίνεται με το χρέος και με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Συγχρόνω όμω δεν πρέπει να αγνοείτε την κοινωνική διάσταση. Τα καλύτερα και τα χειρότερα μα έρχονται από τι ΗΠΑ. Για δείτε πώ έχουν φτιάξει αυτή την οικονομία του. Υπάρχουν ε, αυτοματισμοί. Σας ζητάμε λοιπόν να κάνετε κι εσείς το ίδιο στο κοινωνικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η κρίση έχει και κοινωνικές ε, ε, και κοινωνικούς λόγους, αλλά έχει και κοινωνικές συνέπειες. Η κοινωνική διάσταση λοιπόν πρέπει να βρεθεί στην καρδιά και να υπάρξει ένας αυτόματος σταθεροποιητής βάσει ενός ελάχιστου επιδόματος ανεργία Είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο και είναι αυτό το οποίο θα σας επιτρέψει να διορθώσετε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που δεν καταφέρνετε να ξεπεράσετε με τη δικιά σας πολιτική. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εμείς ήμασταν σε μια κατάσταση κρίσης επίσης σοβαρής όπως η σημερινή και χάρη στο Walter State καταφέραμε να ξεφύγουμε. Σήμερα έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα, αν μας άκουγε ο, Επίτρο, ο Πρόεδρος Επιτροπής των Παρόσο να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο. Και αν θέλετε, η εμβριακή κατάσταση αυτή τη λύση είναι αυτό ακριβώ που σα ζητάμε, οι αυτόματοι σταθεροποιητέ. Με τον Επίτροπο Αντόρ λοιπόν σας ζητάμε να προχωρήσετε στον αυτόματο αυτό σταθεροπιστή έτσι ώστε να έχετε ε, δώσει το κύριο αυτού του συστήματος, τον κύριο το σπόρο να βάλετε για αυτή τη λύση που όλοι περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπερές, το λόγο έχει τώρα η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Υποθέτω ότι αναγνωρίζεται η κέρια σημασία του κοινωνικού πυλώνα στις λέξεις αλλά δυστυχώς όχι ακόμα στις πράξεις. Ο Επίτροπος Άντορ Πέρυσι τον Ιανουάριο μας μίλησε για την κοινωνική διάσταση και είπε ότι είναι απαραίτητη για να νομιμοποιηθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και για να γίνει αποδεκτή η Οικονομική και Νομισματική Ένωση από τους πολίτες. Ε, μόνο αν ενισχυθεί η νομιμοποίηση και η αλληλεγγύη ταυτόχρονα θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Αληθεύει αυτό, όμως δεν έγιναν ταυτόχρονα οι δύο προσπάθειες. Ναι, ακούσαμε πολλά για τη δημοσιονομική πειθαρχία, όμως η νομιμοποίηση και η αλληλεγγύη καταλαβαίνετε πώς ακούγονται στο μυαλό των καταθετών στην Κύπρο των Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή τα εκατομμύρια ανέργων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, καλά τα λόγια. Αλλά τι γίνεται με τις πράξεις. Ε, βλέπω ότι γίνεται και με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης όπου ακόμη υπάρχει η ανασταλτική ε, μειοψηφία στο Συμβούλιο και που αρεμποδίζει την ορθή λειτουργία του Ταμείου. Βλέπουμε τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βλέπω επίσης τι γίνεται με το Ταμείο για τους Απόρους. Πάλι η ίδια ανασταλτική μειοψηφία στο Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταλήξει στην ένδυα και δεν εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Είναι απίστευτο και δεν καταλαβαίνω πώ κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τέτοια προγράμματα διότι ισχυρίζονται ότι συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μα αυτό τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Επίση, αν δούμε τα ηχέγγυα για την νεολαία και πάλι εδώ, διαφωνία για τη συμπερίληψή του στο κοινωνικό Κοινωνικό Ταμείο έχει παραμείνει στο στάδιο σύστασης και μόνο. Τι μήνυμα περνάει αυτό στους νέους, τους άνεργους νέους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα λοιπόν δεν συνεργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων. Επίτροπε, ναι, πολύ ωραία τα λέτε. Μας είπατε ότι χρειαζόμαστε κάτι καινούργιο για να αντιμετωπίσουμε την νεολαία. Δείτε όμως την πράξη τι συμβαίνει. Υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Χαρκίν, κυρία Κορνέλησεν. Τώρα δύο λεπτά παρακαλώ. Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Αντόρ έχει, μας έχει ενθαρρύνει για το τι πρέπει να κάνουμε. Ότι χρειάζεται περισσότερη αλληλεγγύη, μας λέει. Ότι είναι πολύ βασικό αυτό. Βοηθάμε κάποιον για να βοηθήσουμε και το κοινό καλό. Πολύ βασικό αυτό. Τρία χρόνια τώρα προσπαθούμε να επιβάλλουμε δημοσιονομική λιτότητα με οικονομικά μέτρα. Η αλληλεγγύη δυστυχώς έχει ξεχαστεί. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει τώρα ένα νέο σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το Συμβούλιο όμως πρέπει τώρα να ξεκινήσει, όχι αργότερα. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την οικονομική ενοποίηση, αλλά να κοιτάμε και την, κοινωνική διάσταση. Είναι πολύ βασικό αυτό και χαίρομαι που η Επιτροπή επιτέλους το κάνει μετά από το πακέτο των έξι νομοθετικών προτάσεων. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τις κοινωνικές υποθέσεις, γιατί τα χρέη, η ανεργία πνίγουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις γυρνάνε γύρω από την ανταγωνιστικότητα. Κάτι το οποίο όμως έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχύει τις ανισότητες. Φοβάμαι ότι Χρειαζόμαστε κάτι και για την οικονομική ισορροπία με μέτρα, με κυρώσεις κτλ. Τα κράτη-μέλη να μπορούν να βασιστούν σε ένα σχεδιασμό για να προχωρήσουν, αλλά χρειάζεται συγχρόνως και ένα άλλο σκέλος που θα είναι η κοινωνική διάσταση για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αφαίρουν στην Ευρώπη. Χρειάζεται ένας συντονισμός. Περιμένω τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι κοινωνικά μέτρα θα πάρει. Να μην πρόκειται για ένα συμβολικό και μόνο συμβολική χειρονομία, αλλά να πρόκειται για πραγματικά κοινωνικά μέτρα και να υπάρξει και ένα βαθμολόγιο ώστε να δούμε ποιος κάνει τι τελικά για να καταπολεμηθεί η ανεργία και η ένδια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βιζότο έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Τα στοιχεία και τα δεδομένα του Μαρτίου από τη Eurostat είναι σαφέστατα. Υπάρχει ύφεση, συρρήκνωση της οικονομίας. Πρόκειται για την ε, πιο μεγάλη ύφεση από την στιγμή που γεννήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινωνόμισμα. Αυτό που μπορούμε να σώσουμε πρέπει να το διασώσουμε. Είναι όμως κάτι που γίνεται με πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Σήμερα δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, κλείνουν σχολεία, δικαστήρια. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε οι πολίτες να ζουν πραγματικά σε συνθήκες φτώχειας και ένδυας και θα δημιουργήσουμε, αν συνεχίσουμε, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες μία κατάσταση όπου η πλειοψηφία των νέων θα είναι άνεργη και θα οδηγηθούμε σε μια πραγματική τραγωδία. Καθημερινά βλέπουμε αυτοκτονίες στην Ευρώπη. Η πολιτική λιτότητα έχει αποτύχει. Αυτό είναι σαφές. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι εμποδίζεται και η επαναφορά στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να διασφαλίσουμε μία πραγματική κοινωνική πτυχή αυτής της ε, πολιτικής. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές ε, σε νομοθετικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των χωρών. Όσον αφορά λοιπόν την κοινωνική πτυχή, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα που θα οδηγούν σε περισσότερη κοινωνική συλλογή. Η ε, κυρία Ματία, σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχει ένας κοινωνικός πυλώνας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μετά από τις δεκαετίες λειτουργίας του ευρώ, αλλά πρόκειται για τον πυλώνα καταστροφής, κοινωνικής καταστροφής. Προ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσει των κρατών μελών έχουν οικοδομήσει επ' αυτής της πολιτικής, καταστρέφοντας τους μισθούς, τις συντάξεις, υποβαθμίζοντας την κοινωνική προστασία, απομιζώντας τους μισθούς όλων για να χρηματοδοτήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές οδηγώντας όλους σε ανεργία, σε ανισότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία καλούμεθα να αντεπεξέλθουμε και κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη μας μιλάνε για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, αυτό που βλέπουμε στους ε, παχυλούς ε, τίτλους του τύπου, ότι, ε, ότι αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας έτσι περαιτέρω, ότι όλοι καταλήγουν στην ίδια κατάσταση και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σταματήσουν σταματήσουν να ισχυρίζονται ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μοντέλο χωρί του ίδιου πολίτε. Δεν αντέχει άλλο ο λαό. Δεν τα αντέχει άλλο. Και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, διότι ε, θα σημάνει αυτό το τέλο του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Θα το συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστούμε η κυρία Φερέιρα. Τώρα 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ε, το πιο απτό τεκμήριο των ανισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. 62% ε, ε, των νέων στην Ελλάδα είναι άνεργοι, 57% στην ε, Ισπανία, 40% στην Πορτογαλία. Πρόκειται για την κοινωνική καταστροφή και είναι απόρρια των πλημελών πολιτικών που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσης ένας λόγος της συνεχούς επιδείνωσης της εσωτερικής κατάστασης στα κράτη-μέλη για δύο λόγους πρόθεσμα Δεν γίνεται πανισορρόπηση δημοσιονομική όταν υπάρχει αυτή η κοινωνική έκρηξη και διαρκεί η ύφεση και τα δημοσιονομικά ελλείμματα πρόθεσμα. Δεν γίνεται να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα όταν όλοι φεύγουν από την αγορά εργασία και μεταναστεύουν σε άλλε χώρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ο Επίτροπο ε, πότε προτίθεται να παρουσιάσει ενώπιον του Κοινοβουλίου αυτό που υποχρεούται να μα παρουσιάσει ω αποτέλεσμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2012 του τέστην ένα κοινωνικό πυλώνα που θα ανταποκρίνεται και στο σκόρ επιδόσεων ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε μειώσουμε την ανεργία, ε, την κοινωνική ένδυα και να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισορροπίες. Ε, αυτό ε, είναι μονόδρομος για μας και μόνο μέσα από την ανάλυση της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής κατάστασης των κρατών μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό μοντέλο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο με ονομαστικές τιμές και δημοσιονομικές πολιτικές. Επειδή λείπει η κυρία Μπιλμπάου Μπαράντικα, ο κύριος Μπλουμ Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση αυτή. Εδώ μέσα ε, μοιάζει να ε, υποθέτουν ορισμένοι ότι το χρήμα φυτρώνει στα δέντρα. Ακούσαμε για τη φτώχεια, την ανεργία, αλλά παρακαλώ ακούστε με, θα σε εξηγήσω γιατί. Είναι παλαβό το σύστημά μας ε, όσον αφορά την ευημερία και σε επίπεδο εταιριών και την κοινωνική προστασία και σε επίπεδο εταιρεών και σε επίπεδο κρατικό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνουμε απόλυτα υγιείς νέους για να μην εργάζονται και εισάγουμε από την Ανατολική Ευρώπη για να κάνουν τις δουλειές. Τι κάνουμε λοιπόν, δίνουμε λεφτά ε, καταστρέφοντας την οικονομία μας και για να πληρώσουμε όλα αυτά χρειάζεται 20% ΦΠΑ, τρομερή, ε, τρομερά επίπεδα ε, φόρων εισοδήματος και επί των επιχειρήσεων. Πώς θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση μόνο μέσω ανάπτυξης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Εάν δεν πρόκειται για την κοινωνική ασφάλιση, έχουμε τις πολύ υψηλέ αμοιβέ προς όλους τους κολλητούς που έχουν τις, ε, επικεφαλής, ε, τις θέσεις των επικεφαλής των επιχειρήσεων. Έχω γνωστούς που έχουν τεράστια αγροκτήματα που παίρνουν επιδοτήσεις για αυτά τα τεράστια αγροκτήματα και ε, επίσης παίρνουν επιδοτήσεις για να βάλουν και τεράστιες ε, ανεμογεννήτριες ε, στα κτήματά τους. Για το όνομα του Θεού, να σταματήσουν όλα αυτά, να σταματήσει η τρομερή φορολογία, να σταματήσει αυτός ο ρολομανδίας της κοινωνικής πρόνοιας, να κάνουμε τους νέους μας να εργάζονται. Ευχαριστώ κύριε Μπλούμο. Κύριο Τούσα, ένα λεπτό. Η Ένωση βαθιά αντιλαϊκή και εχθρική προ τα συμφέροντα τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων, όπω άλλωστε ολόκληρο το οικοδόμημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί την αιγμή του δόρατο για την ενίσχυση των ευρωνοσιακών μονοπωλιακών ομήλων και τη κερδοφορία του. Ο δίθεν κοινωνικό πυλώνα τη ΩΝΕ είναι ανύπαρκτο, ασυμβίβαστο με τη φύση τη και το χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα στη δουλειά των εργαζομένων μετετράπηκε σε απασχολησιμότητα χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασία ισοπαίδωση τη κοινωνική ασφάλιση με μισθού και συντάξει πείνα είκοσι εκατομμύρια άνεργοι εκατόν εκατομμύρια που ζουν κάτω από τα όρια τη φτώχεια απόλυτη και σχετική εξαθλίωση για του λαού στα κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση. τα σχέδια και οι προτάσει για εμβάθυνση τη ονε δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα αντίθετα βαθαίνουν ακόμη περισσότερο τον αντιδραστικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ένωσης μεγαλώνουν την επιθετικότητα των μονοπωλίων ενάντια στην εργατική τάξη τα λαϊκά στρώματα στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης στους λαούς όλου του κόσμου. τα ιδεολογήματα ότι η ευρωπαϊκή ένωση θα εξασφάλιζε τη λαϊκή ευημερία ότι μπορεί να υπάρξει ο ναι, με διαφορετική δίθεν πιο κοινωνική αρχιτεκτονική ότι η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να μετατραπεί από συμμαχία του κεφαλαίου σε ευρωπαϊκή ένωση των λαών αποδείχθηκαν ιδέα ψέματα εξαπάτηση των λαών. Ευχαριστώ κύριε Τούσα. Ο κύριος ε, Θέρκας, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Με κάθε σεβασμό κύριε Επίτροπε, θέλω να σας πω ότι η παρουσία σας, τα λόγια σας μας ε, προκαλούν τεράστια ανησυχία. Η παρουσία σας, γιατί υπάρχει τέτοια τεράστια κρίση, τουλάχιστον ο πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο αρμόδιος επίτροπος θα έπρεπε να είναι παρόν και όχι ο επίτροπος ε, οικονομίας. Γιατί η κρίση μας οφείλεται στην ανισορροπία που παρατηρούμε λόγω της έλλειψης ε, κοινωνικής διάστασης. Και περιμέναμε προτάσεις, μέτρα, ένα δρομολόγιο, συγκεκριμένες ημερομηνίε που να σας δεσμεύουν, όπως είπαμε στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Και τι είδαμε, ένα δάσος από ε, λόγια και μία έρημο συγκεκριμένων προτάσεων. Βεβαίως, χρειαζόμαστε και το είπα και στον Επιτροπάντορ ξέρω ότι ο Επίτροπο Άντορ έκανε ορισμένε προτάσει, αλλά δεν ενεκρίθησαν από το Συμβούλιο. Θα πρέπει να καταλάβει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι είναι τρομερά κρίσιμη η κατάσταση, είναι δραματική η κατάσταση. Επειδή δεν υπάρχει αυτό ο κοινωνικό πυλώνα, στην ουσία παραβιάζουμε τι συνθήκε, παραβιάζουμε την οικονομική λογική. Χάνουμε ζήτηση, χάνουμε δραστηριότητα. Και όλα αυτά δημιουργούν το τεράστιο δράμα της ε, ανεργίας και την έλλειψη φορολογικών πόρων που εξηγούν και τη δημοσιονομική κρίση των λαών. Καταστρέφουμε το κοινωνικό κεφάλαιο των λαών μας. Μας είπατε ότι υπάρχουν περισσότεροι μετανάστε, μετανάστευση. Όχι. Στην ουσία αιμορραγεί η χώρα μας και όλες οι άλλες χώρες όσα, λόγω αυτής της αναγκαστικής μετανάστευσης. Η κατάσταση φαίνεται πως δεν σας είναι κατανοητή πολλαπλασιάζεται τα προβλήματα, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο κοινωνικό αλλά και πολιτικό. Χρειαζόμαστε δείκτε για την κατάσταση όπου είμαστε. Χρειαζόμαστε πολιτική, κοινωνική διακυβέρνηση όπω και οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει οπωσδήποτε όλε ε, οι σημαντικέ ε, συζητήσει να αφορούν και τα κοινωνικά θέματα, όχι μόνο τα οικονομικά. χωρί κοινωνικό διάλογο δεν θα υπάρξει η αναγκαία σωστή πολιτική. Χρειαζόμαστε πολλαπλασιαστέ άλλου είδου. Χρειαζόμαστε ε, αυτόματους σταθεροποιητές. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα για το μέλλον όπου το κοινωνικό να γίνεται σεβαστό από τις συνθήκες όσο και το οικονομικό και οι άνθρωποι να μετράνε όσο η οικονομία και τα χρηματιστήρια. Ευχαριστώ. Κοφεράτη ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η μακρά κρίση την οποία διανύουμε μας ε, αναθέτει τα εξή δύο προβλήματα. Καταρχήν, ε, τη διαρκής μείωση της απασχόλησης και άρα αύξηση της ανεργίας. Έπειτα, διαρκής αύξηση της φτώχειας. Ε, διαρκώς περισσότερα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι αυξήθηκαν πάρα πολύ. Έχουν γίνει δράσεις από πλευράς κομισιών για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Όμως, όσον αφορά την ανάκαμψη και την απασχόληση. Υπάρχει μόνο βασική οδός, η βασική λεωφόρος, αλλά δυστυχώς ε, λεπτομερή μέτρα δεν ελήφθησαν ποτέ. Και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική για την οποία μιλάμε σήμερα το πρωί, ε, χρειάζονται πιο συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ανθρώπων που αναζητούν θέση αλλά δεν βρίσκουν. Ε, η απασχόληση και η συνοχή είναι βασικός παράγοντας για την ανάκαμψη. Διαφορετικά θα υπάρξει διάλυση και δεν θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον. Ελπίζω πως θα υπάρξει μια γρήγορη αντιστροφή τάση για την οποία δυστυχώς σήμερα το πρωί δεν είδα καν ίχνη. Η κυρία Ρέγνερ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα το πω ξεκάθαρα, χρειαζόμαστε αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα. Τώρα, τέρμα. Γεγονός είναι πως ε, η χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απομακρύνονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Οι πλούσιες γίνονται πλουσιότερες και οι φτωχές γίνονται φτωχότερες. Κύριε Επίτροπε, είναι καλό το ότι συζητάτε μαζί μας σήμερα, αλλά καλό θα ήταν να είναι εδώ πέρα και ο αρμόδιος για τα κοινωνικά. Και οι υπουργοί αρμόδιοι για τα κοινωνικά πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την υπόθεση και να μην λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις οι υπουργοί του ΕΚΟΦΗΝ. Και είναι κρίμα που δεν είναι εδώ πέρα σήμερα το Συμβούλιο. Τα δε κοινωνικά είναι ένα ζήτημα επενδύσεων και δεν γίνονται αρκετά πράγματα. Τέλος, δεν χρειάζεται καμία επανάσταση, απλά πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας και να γίνουμε πραγματικά μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Ταρντένι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως και άλλοι, θεωρώ πως αυτό το θέμα του κοινωνικού διαλόγου με χαροποιεί που βρίσκεται στην, στην ημερήσια διάταξη. Είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική της Ένωσης και για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους πολίτες μεγαλύτερη ελεγγύη. Αυτές οι πολιτικές αυτή η πολιτική θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλούς άξονες εργασίας, όπως ε, τα κοινωνικά μήνυμα στην Ευρώπη. Τα απαιτούμε εδώ και χρόνια και κυρίως ένα ελάχιστο εισόδημα που ήδη ζήτησα στην έκθεσή μου για την ε, ε, καταπολέμηση της στόχιας πριν από τρία έτη. Ε, ένα μίνιμουμ δαπανών, ένα μίνιμουμ μισθών, ιδιαίτερα στη Γερμανία, που τις, θέμα που θίγω στις ερωτήσεις που έχω απευθύνει προς τον Επίτροπο Αντόρο, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η Κομισιόν και το Συμβούλιο συνήθως παίρνουν παίρνουν χρόνο μέχρι να κατανοήσουν πως το Κοινοβούλιο έχει δίκιο, αλλά πόσο χρόνο ακόμα χρειάζεται ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να γίνει πιο κοινωνική και αλληλεγγύη. Ο κύριος Γκουτιέρες Πριέτο, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, στην αρχή της συζήτηση είπατε ότι η Επιτροπή καταλαβαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στο κοινωνικό τομέα. Αλλά από ποιον το ζητάτε αυτό, από το Κοινοβούλιο μας, όχι βέβαια. Η Επιτροπή δεν έχει συνέστηση ούτε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που ζούμε, ούτε πόσο αναγκαία φιλόδοξη πρέπει να είναι η πολιτική τη που ζητούν οι πολίτε δηλαδή για να βγούμε από την κρίση. Δεν έχετε συνέστηση τι συμβαίνει στον δρόμο. Μιλάτε για μια οικονομική στρατηγική που είναι απόλυτα αντίθετη σε αυτή που χρειάζεται η Ευρώπη. Θα προκαλέσει περισσότερη ύφεση. Θα αυξήσει τι κοινωνικέ αντιθέσει μεταξύ των πολιτών. Διότι όλα αυτά που λέτε όλα αυτά που λέτε για οικονομική ε, διακυβέρνηση, λέγοντας ότι όλα αυτά θα ε, μας βγάλουν από την κρίση, δεν μας οδηγούν στην επίλυση της κοινωνικής διάστασης. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική ένωση. Αυτή πρέπει να είναι η πολιτική. Ήταν πολύ απογοητευτικά αυτά που μας είπατε. Το Κοινοβούλιο δεν αποδέχεται να συνεχίσει αυτή η πολιτική μόνο βούρδουλα και καθόλου λουκούμι. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε περισσότερα αν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση για την κοινωνική πολιτική, για τους σταθεροποιητές, τους αυτόματους σταθεροποιητές, για την ασφάλεια, για την ανεργία, για ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας. Ανοίξτε τώρα αυτή τη συζήτηση. Πρέπει οπωσδήποτε να ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση. Θα πέσουμε στην άβυσο αλλιώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κουτιέρεθ, λέει πρόεδρος. Μπιλμπάο Μαραντίκα, 1,5 λεπτό. Και μετά θα αρχίσει η διαδικασία προσέλκυση προσοχή του Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο τη ταυτότητά μα. Πρέπει είναι ένα τρόπο να εργαζόμαστε, να προωθούμεθα που αποτελεί σημείο αναφορά σε όλο τον κόσμο. Η Ευρώπη σημαίνει ανάπτυξη αλλά με αξίε. Πρέπει να αφορά τα άτομα το ευρωπαϊκό πρότυπο. Γι' αυτό η κοινωνική συνοχή μαζί με την αηφορία ή και την ε, γνώση είναι το τρίδημο που θα μας επιτρέψει να, να είμαστε ανταγωνιστικοί στον πλανήτη. Πρέπει να έχουμε μια τέτοια πολιτική, ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό dumping και την ε, κερδοσκοπία. Η εικόνα που έχουμε τώρα της Ευρώπης είναι ε, λιτότητα και περικοπές. Πρέπει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, να βελτιωθεί η εφαρμογή των δικαιωμάτων ανθρώπων. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα επιτύχει μόνο εάν έχει ανθρώπινη διάσταση, αλληλεγγύη, εμπιστοσύνη, απασχόληση, αναγνώριση και σεβασμός για όλους, με κοινές προδιαγραφές και κοινά όργανα που να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις μαζί με την πολυμορφία που χρειάζεται και να αξιοποιήσουμε όλη την αναγκαία γνώση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες μας τις γνώσεις και κύριε Επίτροπε σας παρακαλώ να αξιοποιήσετε τα πιο αναγκαία εργαλεία αλλά μην ξεχνάτε τους ανθρώπους, τους πολίτες που υποφέρουν από τόσα δεινά σε αυτή τη συγκυρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχή ε, της Προέδρου. Η κυρία Ζαζοβιέφκα, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μέχρι στιγμή στη συζήτηση για την κρίση η κοινωνική πτυχή δεν είχε συζητηθεί γιατί τα επίγοντα ήταν τα οικονομικά. Εστιάσαμε στην πρόληψη της ε, κρίσης και ε, βέβαια καταλήξαμε σε αυτό το οποίο βλέπουμε στην Ελλάδα και την Ισπανία. Ε, θα πρέπει λοιπόν η ΟΝΕ να συμπληρωθεί με κοινωνικές επενδύσεις. Αυτό είναι σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, για να ξανάρθει η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες πρέπει να πάνε χέρι-χέρι με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για κοινωνικές επένδυσεις επιπλέον. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί κοινωνικός έλεγχος όπως έχουμε ελέγχου στην οικονομία έτσι ώστε ε, να παρακολουθούμε καλύτερα τις δραστηριότητες ε, των κρατών μελών. Δεύτερον, δεν θα υπάρξει πραγματική ένωση χωρίς κοινωνική σύγκληση. Αυτό το οποίο ήταν το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα έχει μετατραπεί σε κοινωνικό ντάμπινγκ. Αν είναι να υπάρχει κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να αναπτυχθούν τα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμα, έτσι θα έχουμε και καλύτερη κοινωνική σύγκληση. Σας ευχαριστώ κυρία -Κάστα. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος ο κύριος Ρέν εξακολουθεί να θέλει να ακολουθήσει την ίδια πορεία λιτότητας για όλους. Κάτι το οποίο βέβαια αρνείται και τα πραγματικά αποτελέσματα. Οπότε δεν υπάρχει νομίζω πλέον καμία λογική για την λιτότητα και υπάρχουν τεράστια, πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας. Και έτσι βεβαίως δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να γίνεται και ακόμη χειρότερο το δημόσιο χρέος. Δεν ξέρω λοιπόν, κύρια Πρέντεργκαστ, λίγο πιο σιγά αν μπορείτε, γιατί δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. το μέσο ανταγωνιστικότητας που βασίζεται σε διμερείς συμβάσεις μεταξύ κομισιών και κρατών μελών θα βραχικυκλώσει τη δημοκρατική λογοδοσία και θα αγνοήσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Θεωρώ πως συμβάσεις αυτές θα γίνουν κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να μειώσουν τους μισθούς, να καταπατήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να επιβάλλουν περαιτέρω περικοπές στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Ένα κοινωνικό σύστημα για την ΟΝΕ θα πρέπει να έχει και τους κατάλληλους πόρους για να αντισταθμίσει τις ανισορροπίες της Ευρωζώνης. Οπωσδήποτε λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική διακυβέρνηση ε, χωρίς αλληλεγγύη. Και δεν είναι δυνατόν να κρυβόμαστε πίσω από το φύλλο των περικοπών. Σας... Η κυρία Σοπάσκα, ευχαριστώ. Κύριο Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση κυρίαρχων κρατών που δημιουργήσαν μια συντονισμένη πολιτική και οικονομική ε, βάση με βάση μια ε, συνθήκη. Τα μέσα που προτείνει η Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση πρέπει να σέβονται αυτή τη βασική αρχή και δεν θα πρέπει να περιορίζουν τη δυνατότητα των κρατών και κυβερνήσεων και κοινοβουλίων να καθορίζουν την οικονομική και κοινωνική του πολιτική. Τα περισσότερα, τα περαιτέρω βήματα για την οικονομική και δημοσιονομική ένωση που προτείνει ο Γάλλο πρόεδρο δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρί να αλλάξει η συνθήκη τη Λισαβόνα, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι οι πολίτε μα θα πρέπει να το αποδεχθούν. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό σχέδιο καταραίει σε όλε τι χώρε και οι πολίτες όλο και περισσότερο θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις τους, τα κοινοβόλια τους είναι πιο αρμόδια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Αυτή η προσπάθεια συγκέντρωσης εξουσιών στο κέντρο δεν συνάδει με αυτά που πιστεύουν οι πολίτες μας. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να ε, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε περισσότερη εναρμόνιση και συνεργασία και όχι μεταβίβαση αξιοδιοτήτων. Ευχαριστώ η κυρία Κάντεμπακ. Κυρία Πρόεδρε, λάβαμε το βραβείο ειρήνης ε, πρόσφατα και όχι μόνο για αυτά που επιτύχαμε στο παρελθόν, αλλά και για όσα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Και η ειρήνη είναι και κοινωνική ειρήνη, η κοινωνική συνεργασία και Έχετε δώσει απαντήσει σε αυτέ τι ερωτήσει, παρακαλώ. Έχουμε, για παράδειγμα, λάβει ένα κείμενο που λέει να επενδύσουμε στην υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλέ συστάσει που θα επέτρεπαν να αναπτυχθεί η κοινωνική Ευρώπη. Θα επέτρεπαν επενδύσει στον τομέα τη υγεία, επενδύσει στην υγεία των ανθρώπων, επενδύσει στην εργασιακή υγεία, επενδύσει στην οικονομία, στην ε, κοινωνική συνοχή αλλά αυτό που κάνετε κάθε μέρα είναι στην ουσία το αντίθετο με όλες τις θαυμάσιες ε, προτάσεις που έχετε κάνει. Καλείτε τα κράτη να κάνουν περικοπές στον τομέα της υγείας αντί μέσω πραγματικών προγραμμάτων να ε, τους ε, ενθαρρύνετε να επενδύουν στον τομέα αυτό της υγείας, της υγείας των ανθρώπων, της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχει λοιπόν κείμενο με προτάσεις, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση να τις εφαρμόσετε. Ευχαριστώ και η κυρία Γιάκον Σάριν τώρα τελευταία στη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν πρόκειται να διατηρηθεί η ΟΝΕ να λάβουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση. Ακούσαμε πως ε, μέχρι στιγμής ε, δεν βλέπουμε να λαμβάνεται υπόψη σωστά η κοινωνική διάσταση. Προφανώς η ανταγωνιστικότητά μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ικανότητά μας να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο και να παραμείνει ο κόσμος στην αγορά εργασίας. Όσο περισσότεροι βγαίνουν εκτός αγοράς εργασίας αυξάνεται το χρέος μας και πέφτει η αξιοπιστία μας. Ε, θεωρώ λοιπόν πως η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και ο Επίτροπος θέλουν ε, μια πιο δημοκρατική και δικαιότερη Ευρώπη και μια κοινωνικά βιώσιμη Ευρώπη. Υπάρχει νομίζω ένταση μεταξύ των διαφορετικών αυτών σκοπών και καλό είναι να προωθήσουμε την κοινωνική διάσταση της ΩΝΕΣ. Σας ευχαριστώ κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι βουλευτές, μου ζήτησε ο πρόεδρος Μπαρόζο και ο επίτροπος Άντορ να ε, παραβρεθώ σε αυτή την συζήτηση. Άλλαξα το πρόγραμμά μου και διάφορες υποχρεώσεις στις ε, Βρυξέλλες που αφορούσαν τις συστάσεις αναχώρα της επόμενης εβδομάδας γιατί αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της απασχόλησης και στα κοινωνικά θέματα και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Να σχολιάσω κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Ξεκινώντας την κυρία Κορνέλισεν που αναφέρθηκε στον πίνακα βαθμολογίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης στην οικονομική διακυβέρνηση. Κατά την άποψή μου υπάρχει περιθώριο για να ληφθεί υπόψη ε, η κοινωνική διάσταση στα υφιστάμενα εργαλεία που έχουμε. Παραδείγματο χάρη, ένα πίνακα βαθμολογία απασχόληση και κοινωνικών δικτών με βάση τα υπάρχοντα μέσα θα βοηθούσε να ανοιχνεύσουμε καταστάσεις ε, κοινωνικών εντάσεων και ανισορροπιών και να οδηγηθούμε σε γρήγορες ε, διορθωτικές ενέργειες. Η εποπτεία αυτή θα βοηθήσει πρώτα απ' όλα στο να δώσουμε έμφαση στην διάσταση της κοινωνικής πολιτικής όταν λαμβάνουμε μακροοικονομικές αποφάσεις στο επίπεδο Ευρώπης και κρατών μελών και δεύτερον να ενισχύσει την παρακολούθηση κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών αποσχόλησης για να μπλύνουμε τις συνέπειες άλλων πολιτικών. Νομίζω πως έχουμε πολλά να δεχτούμε ένας από τον άλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών ήδη λαμβάνει η χώρα στους ε, μηχανισμούς ε, κοινωνικού συντονισμού και έτσι θα μπορούμε καλύτερα να συντονίσουμε τον εξάντε συντονισμό. Επίσης η κοινωνική διάσταση μπορεί επίσης να ε, φαίνεται και στο μέσο σύγκλησης. Αρκεί να υπάρχει και μια στήριξη οικονομική, η οποία θα διευκολύνει την εφαρμογή τέτοιων μέτρων, παράδειγμα χάρη ένα κράτος μέλος το οποίο θα δεσμεύεται να εφαρμόσει δύσκολες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορεί να λαμβάνει ε, χρηματοδότηση για προγράμματα διαβίου κατάρτισης για να βελτιώσει την απασχολησιμότητα των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων. Αναφερθήκατε επίσης στους κοινωνικούς εταίρους. Εξυπακούεται πως η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ αφορά και την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων ε, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αποδεχθούν αυτές οι πολιτικές ε, και να ενισχυθεί έτσι η Ευρωζώνη. Η εμπλοκή και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους στο εθνικό επίπεδο είναι βεβαίως κέρια σημασίας και πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω. Και αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις πως πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να καταπολεμήσουμε την κρίση της ανεργίας και ειδικά της ανεργίας των νέων. Και γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, ειδικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Εδώ πέρα έχουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για την Νεολαία, που βασίζεται στις εμπειρίες και τα αποτελέσματα πύχη των σκανδιναβικών χωρών και δίνει στους νέους την ευκαιρία να έχουν είτε μια θέση εργασίας, είτε κατάρτισης, είτε εκπαίδευσης και έτσι βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους και τους βοηθάει όταν θα επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, όταν θα μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση. Ε, κατά την άποψή μου, αυτή είναι μία από τις ε, βέλτιστες ε, πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω πως μπορούμε να επεκτείνουμε αυτή την εγγύηση για την νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, να επισημανώ πως για το επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο που έχουμε προτείνει λέμε πως 25% της ε, χρηματοδότησης συνοχής πρέπει να πάει στο κοινωνικό ταμείο και το ίδιο το κοινωνικό ταμείο θα αυξηθεί η χρηματοδότησή του κατά 10%, 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Καθήκον του είναι να αυξήσει τις δυνατότητες απασχόλησης, ε, να παρέχει κατάρτιση και διαβίου εκπαίδευση να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη και να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Επιπλέον, έχει προταθεί τουλάχιστον 20% συνολικών πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε κάθε χώρα να πηγαίνουν για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, Τώρα θα πατήσω στα φιλανδικά στην κυρία Γιακονσάρη γιατί ε, ε, ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Είπε πως δεν πρέπει να θεωρούμε πως η κοινωνική και η οικονομική πτυχή είναι αντιφατικές. Και εγώ συμφωνώ, το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο ότι έχουμε αποτελεσματική οικονομία και παράγουμε θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα φροντίζουμε και τους πιο αδύναμους. Για να μπουν στο αγορά εργασίας. Και οι δύο διαστάσεις πρέπει λαμβάνονται υπόψη και η κοινωνική διάσταση στην ΩΝΕ είναι πάρα πολύ σημαντική και η Κομισιόν θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Οπότε κλείνει η συζήτηση. για το θέμα αυτό, οπότε διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 12 που θα αρχίσουν ψηφοφορίες.